Please can we adopt the agenda? Να συνεχίσουμε την ημερησία διάταξη. Σας μεθυμίζω ότι μεταδίδεται στο ίντερνετ η συνεδρίαση. Και έχετε και το καινούργιο ενημερωτικό δελτίο και έχουμε και την εφαρμογη e-meeting. Επίσης, σας θυμίζω ότι θα έχουμε στις 30 Μαΐου έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τρεις με εξήμιση. Um, Γράψτε το και σημειώστε το. Επίσης, ε, αν θέλετε μπορείτε να βρείτε και το σημείωμα πρακτικών σε σχέση με την ε, ομάδα εργασίας για την πνευματική ιδιοκτησία. στο βάθος τη αιθούση, δίπλα στις ε, εισόδου τη αιθούση και όποιος ε, θέλει μπορεί να λάβει και άλλα αντίτυπα ή αν δεν Ας εγκρίνουμε τα πρακτικά θέλουν εγκεκριμένα δεν υπάρχει ένα με το συνεδρίαση και τώρα συνεχίζουμε όσον αφορά τα εικονικά νομίσματα. Είναι μια γνωμοδότηση και η συγκητή είναι η Λουρίκε Τρεμπέσιου. Λουρίκε, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες λοιπόν να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Όλοι οι ομάδες υπέβαλαν ε, ενδιαφέρουσες προτάσεις, αντικειμενικές και έδειξαν ε, επικοδομητική διά, διάθεση. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Το έγγραφο το οποίο συγκέντρωσε μεγάλη υποστηρίξη είναι ε, πολύ τεχνολογικά και υπέρ της τεχνολογίας. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να κρατήσουμε ε, την θέση μας σε ό,τι αφορά την τεχνολογική κοινοτομία. Οι εικονικές εξελίξεις είναι μεγάλες ε, εξελίξεις, γιατί ως τώρα ήταν σαφές προς τα που θα κινηθούν οι τεχνολογίες. Και για τον λόγο λοιπόν αυτό θέλουμε να αποφύγουμε την ρύθμιση και αυτές οι προσεγγίσεις θα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία ανάπτυξης και θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα και για, άλλες, ε, ε, για άλλους κλάδους. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με εικονικά νομίσματα, ε, είναι δύσκολο συχνά να παρακολουθούν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικές ε, δραστηριότητες και για τρομοκρατία. Αλλά σε ό,τι αφορά το ρευστό χρήμα, υπάρχει ακριβώς η κατάσταση και θέλουμε λοιπόν να μείνει έτσι η κατάσταση αυτή, γιατί ε, είναι και ταυτόσημη της ελευθερίας κινήσεων. Έχουμε λοιπόν ε, θεματική οργάνωση των ζητημάτων αυτών και ελπίζουμε να τα ψηφίσουμε αν μπλοκ. τώρα δεν υπάρχουν ε, σημαντικές ενδείξεις ότι θα προκύψουν και θα ανακύψουν αυτές οι δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν συμπεριλάβαμε την πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει μια task force ε, και να επεκτείνει ενδεχόμενη task force ό,τι αφορά το ξέπλυμα του χρήματο και την τρομοκρατία. Πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα. Ακολουθήσαμε την πρόταση του ΕΛΚ και καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις ε, φάσεις ε, σύνδεσης μεταξύ εικονικών και πραγματικών νομισμάτων να ακολουθήσουμε τα διεθνή πρότυπα. Σοσιαλιστές και δημοκράτες πρότειναν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία να επεκταθεί στην πλατφόρμα αυτή και το συμπεριλάβαμε ως πρόταση σε ό,τι αφορά την εκτεταμένη ρύθμιση. Πιστεύω ότι είναι αρκετά πρόημο το στάδιο αυτό. Καταρχάς δεν θέλουμε να περιορίσουμε την ε, δημιουργικότητα και θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα να δοκιμαστούν διάφορες μέθοδοι. Πρώτη να εγγυηθούμε την διαφάνεια για τον χρήστη, αλλά στην τελική ανάλυση θα πρέπει ο χρήστη να μπορεί να αποφασίζει ποια προϊόντα θα ήθελε να χρησιμοποιήσει. Θεωρώ ότι ο πολίτης είναι σωστά ενημερωμένος για να μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καταναλωτής να μπορεί να κατανοεί τους κινδύνους και τις δυνατότητες. Και κάτι με τη σχετική γραμμή του ΕΛΚ που υποστήριξε ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Δύο καλές τροπολογίες, η 8 του ΕΛΚ και η 39 των Πρασίνων, δεν τη συμπεριέλαβα και έβαλα και αρνητικό πρόσημο στον κατάλογο των ψηφοφορίας. Και αυτό γιατί Θέλω να προαγάγω την τεχνολογική ουδετερότητα. Αυτό υποστηρίχθηκε και από την άλλη στο παρελθόν και θα ήθελα να συνεχίσω το πνεύμα αυτό και βλέπουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία DIT είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ως τεχνολογία αλλά με θέματα αποθήκευσης και εξίσωσης των δεδομένων δεν θεωρείται θετική από όλους τους φορείς. Ενδεχομένως στο τέλος τελικά να επικρατήσουν άλλες τεχνολογίες, λιγότερο τεχνολογικά πολύπλοκες. Θα ήθελα να υποστηρίξω την εξέλιξη του DLT, αλλά να μην αποτελεί τη μοναδική βάση για τα εικονικά νομίσματα. Και για να τονίσω πόσο υποστηρίζω τα ζητήματα αυτά, η ΕΝΕΑ θα την υποστηρίξω των σοσιαλιστών κατά την ψηφοφορία σε ό,τι αφορά ε, την ανεξαρτησία της τεχνολογίας. Ε, κατά τα άλλα, ζητούμε οι stakeholders, για παράδειγμα, οι μπλεκόμενοι φορείς ε, στα πανεπιστήμια να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή στο μέλλον. Για το DLT υπάρχουν, για παράδειγμα, ενδιαφέρουσες προοπτικές σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία και την ε, συναλλαγές σε ό,τι αφορά τα αξιόγραφα, τα κίνητα και το καθεξής. Και τέλος θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για την καλή συνεργασία και ελπίζω η αυριανή ψηφοφορία να μπορέσουμε να τη θεωρήσουμε όλοι επιτυχή. Η γραμμή μας ελπίζουμε δεν αληθεί υπόψη και από την Καθηλή Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια, κύριε Τρεπέσιου. Συντώνησε τη συζήτηση με του κοιόδης εξαιρετικά, με εξαιρετικό τρόπο. Και πάντοτε ε, άκουγε προσεκτικά τις διάφορες ε, προτάσεις των πολιτικών ομάδων με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη και πλήρη έκθεση που αναδεικνύει και τα πλεονεκτήματα και κάποιους από τους κινδύνους των εικονικών νομισμάτων. Στην Επιτροπή αυτή ε, το ζητούμενο είναι να αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες, αλλά και τους πιθανούς κινδύνους. Τα εικονικά νομίσματα είναι μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει σε, να γίνονται γρήγορα συναλλαγές με αποκεντρωμένο τρόπο και σε γενικές γραμμές ασφαλής. Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού των συναλλαγών. αλλά δεν είναι πάντα σαφές πόσο, ποιος είναι ο βαθμός ασφαλείας αυτών των συναλλαγών. Η τεχνολογία του, κατά, του νομισμάτων κατανεμημένου καθολικού και γενικά των οικονομικών, νο, ε, ε, νομισμάτων χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, κυρίως σε διασυνοριακές συναλλαγές δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών Αυτό είναι επιθυμητό για λόγους ανταγωνιστικότητας. Επομένως με τη χρήση των εικονικών νομισμάτων αμέσως εταιρεία που τα χρησιμοποιεί γίνεται πιο ανταγωνιστική. Αλλά βέβαια υπάρχουν και κίνδυνοι με τα, με τα εικονικά νομίσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως η τρομοκρατία ή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να, να δημιουργήσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως να υπερβάλλουμε. Δεν θέλουμε να καταπνίξουμε αυτή τη νέα τεχνολογία και την καινοτομία με τους κανόνες μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα χρησιμοποιηθεί και πού θα φανεί χρήσιμη η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού. Γι' αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε θα φανει χρησιμη η τεχνολογια νεμιμενου καθολικου αρκετά ε, ευέλικτο, αρκετά ευρύ. Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούν και με τις θέσεις του ΕΛΚ. Επομένως, συνολικά θα υποστηρίξουμε την εκθέση αυτή. Ευχαριστώ. Ντάντη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα, Πρόεδρε, ευχαριστούμε την εισηγητρία για τις προσπάθειές της και τους συνεργάτες της αλλά και τους άλλους χιώδεις γιατί αυτό το οποίο σήμερα θα προκύψει αύριο θα οδηγήσει σε έγκριση των τροπολογιών και έτσι θα έχουμε μια επιτυχία στο μέτωπο ενός ακαθόδου θέματος που ε, θα έχουμε κάποια θετικά στοιχεία και βέβαια όπως ε, για όλα ε, υπάρχει και κάποιο ρίσκο πάντως θεωρώ ότι είναι η έκθεση με αυτές τις Συμβασικέ τροπολογίες με τις οποίες εμείς συμφωνούμε. Ε, καλύφθηκαν ε, όλες οι έννοιες μας, οπότε αισθανόμαστε καλυμμένοι και έχουμε εδώ πέρα τα εξή δύο στοιχεία, το ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθηθεί αυτή η σημαντική νέα τεχνολογία, ούτω ώστε να αποσπάσουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, κάποιες ευκαιρίες ε, και όχι μόνο για τον κλάδο του οικονομικού την μεριά ε, είναι και θέμα της ύλης της δικής μας ε, επιτροπής γιατί θα πρέπει να προσφέρουμε κάποιες εγγύησεις στους ε, καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν τα οικονομικά, τα οικονομικά νομίσματα και έτσι να έχουν ταυτόχρονα κατοχυρώσει και τα χρήματά τους. Για να σταθώ τώρα σε κάποια σημεία που επισημάναμε και θέλουμε να τα τονίσουμε. Πρώτα πρώτα μιλάμε για μια προσέγγιση ευρωπαϊκή, κοινή και χρειάζεται επομένω συντονισμός ε, οριζόντιος για το θέμα αυτό και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήριες ούτως ώστε να είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής. Υπάρχει εδώ συμβαστική τροπολογία γιατί είναι σημαντικό το θέμα για μας επίσης το πώς θα ε, συγκροτηθεί μια task force και αυτή θα μπορέσει να αναλύσει την εξέλιξη ε, αυτού του καινοτόμου συστήματος του εικονικού νομίσματος και κυρίως όσον αφορά τις τεχνολογίες blockchain ούτως ώστε ε, όλοι να ωφεληθούν παντού όπου θα εφαρμοστεί ε, το εικονικό νόμισμα. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι δυνάμοι τα είπε και η, ε, κυρία Πέλς, τα είπε και η συγκήτρια. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραπέμπουμε για το κοινωνικό σε κάποιο συγκεκριμένο διεθνή πρότυπα. Και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει κατά πόσο και η ε, οδηγία για τη διάθεση προϊόντων εγκλήματος να καλύψει και τα οικονομικά νομίσματα. Έχουμε και εδώ πέρα μια τροπολογία επίσης, Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να φρενάρουμε την καινούργια τεχνολογία, το blockchain και νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα ενδυνάμει πλεονεκτήματα από κάποιε χρηματοοικονομικές υπηρεσίε που θα προκύψουν έτσι. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτική ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη και έτσι να προσθέσουμε καταναλωτή και να βοηθήσουμε εύρυθμη λειτουργία της ενιαία αγοράς. Ευχαριστώ του και την ε, ε συντακτή του κειμένου. Νομίζω ότι θα προκύψει ένα ε, χρήσιμο κείμενο με τις τροπολογίες για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά και λεπτό. Ο επόμενο. Εδώ έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα καινοτομία. Δεν έχουμε ενδιάμεσους, γίνονται όλα πιο γρήγορα. Αν κάποιο στείλει ένα έμβρισμα, παίρνει κάποιε μέρε, κρατάει ε, ενδιάμεσα τράπεζα λεφτά, ενώ όλα γίνονται ακαριέα με το εικονικό νόμισμα. Θα υποφεληθούν όλοι στην Ευρώπη, ο κύριο Γκόγκα Και θεωρώ την μπορεί να υπάρξει ασφάλεια, θα πρέπει να ξέρει πώ θα χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία. Φαντάζομαι ότι bitcoin δεν έχει κανένα από του πολιτικού. Προσπαθούμε δηλαδή να νομοθετήσουμε για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό προτείνω όλοι να αποκτήσετε κάποια bitcoins και έτσι να μάθετε το σύστημα γιατί πρόκειται για την εξέλιξη, πρόκειται για ένα μεγάλο άλμα προς την εμπρός και μεγάλη ευκαιρία. Και το μεγαλύτερο ρίσκο είναι εμείς να είμαστε συντηρητικοί να φρενάρουμε αυτή την εξέλιξη και την έρευνα. Ε, ε, είχε αναπτυχθεί μεγάλη δραστηριότητα σχετικά με αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα, ε, πρώτη για αυτή την τεχνολογία blockchain. Και η εξέλιξη γίνεται με άλματα και ταχαίως. Όλοι προτείνω. να δείξετε θετική στάση και να ψηφίσετε το κείμενο. Βεβαίω είπαμε ότι μπορεί να βοηθήσει οι κλιματικέ δραστηριότητε, ότι υπάρχουν κάποια κίνδυνοι για του ε, καταναλωτέ. Ε, ε, εντάξει, αυτά όλα τα λέμε, αλλά δεν υπάρχουν ε, ενδείξει και στοιχεία. Είναι τόσο μικρό ο κίνδυνο που δεν νομίζω θα πρέπει να φρενάρουμε αυτή την τεχνολογία. Α εξελιχθεί η τεχνολογία και όταν εξελιχθεί, όταν μεγαλώσει, και αποδίδει, τότε να δούμε πώς θα την ε, ρυθμίσουμε ακόμη περισσότερο. Επίσης θα πρέπει να μπορεί να ανοιχνευθούν οι, οι, συναλλαγές. Μα ε, επιδέχονται αυτά τα εικονικά νομίσματα την ανοίχνευση ε, και όχι τα, ε, τα, τα, μετρητά. Άρα σε αυτή τη φάση ας πράσινο φως. Και ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκουόγκ. Ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μας ότι οι συμβαστικές τροπολογίες κινούνται προς σωστή κατεύθυνση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη, τη συνειδητοποίηση και την ευαισθητοποίηση του πολίτη και του καταναλωτή και τη διαφάνεια. Μπορεί να ήταν χρήσιμο να γίνει αναφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τις τροπολογίες ως έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ούλρικε, θες να δευτερολογήσεις. Ναι, και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους κοιόντες εισηγητές, όλους τους ε, βοηθού και υπαλλήλου που μα βοήθησαν για την κατάρτιση τη έκθεση και το ακούσαμε ήδη ότι ήταν καλή η λύση που βρήκαμε για ένα δύσκολο ζήτημα και νομίζω ότι τελικά είναι ισορροπημένη η έκθεση. Δεν θέλουμε ούτε να δώσουμε ελεύθερο πεδίο στην οργανωμένο εγκλήμα, ούτε όμως να καταλήξουμε σε υπερβολική ρύθμιση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την επικοδομητική συνεργασία. Η Πρόεδρος. Θα αλλάξουμε θέσεις τώρα γιατί ο κύριος Ντάντη θα προεδρεύσει τις υπόλοιπες συνεδρίασεις της Επιτροπής. Η επόμενη συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για την οδηγία των προβόλων όπλων και είμαι εγώ η συγγήτρια και θα δώσω λοιπόν τα είναι της τις στον κύριο Ντάντε για να μπορέσω να συγκεντρωθώ. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori, eh, siamo al eh, punto 6 dell'ordine del giorno, controllo dell'acquisizione del possesso delle armi. Μάλιστα, eh. είμαστε στο σημείο 6 τη ημερησία διάταξη σε ό,τι αφορά τα πυροβολά όπλα και θα δώσουμε το λόγο πάρα αυτά στην εισηγητρία, στην κυρία Φόρντ. Thank you. I know that there is a huge... Σας ευχαριστώ. Είναι γνωστό ότι το θέμα αυτό ε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε λάβει email, προτάσεις από ε, πολλού πολλούς ανθρώπους εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ευχαριστούμε όλους για τις προτάσεις τους. Αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο εξτάζεται από τα δικαστήρια μια υπόθεση για 30 πυροβόλα όπλα που βρέθηκαν τα οποία θεωρητικά ήταν απενεργοποιημένα, αλλά στην πράξη εύκολα μπορούσε κανείς να τα απενεργοποιήσει. Τα πέρασαν λαθρέα από τη μάχη και αν κάποιος τρομοκράτης τα είχε ε, αποκτήσει, θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε στο Λονδίνο μια επίθεση αντίστοιχη με εκείνο το που έγινε στο Παρίσι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα και υπάρχουν παρεθυράκια στην νομοθεσία. Η νομοθεσία που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα όπλα που τα πενεργοποιημένα ε, είναι από το 1991 και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας υπέβαλαν τροπολογίες με διάφορες προτάσεις και βεβαίω θα συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ τροπολογίε και κάποια πράγματα φυσικά θα τεθούν και σε ψηφοφορία. Όσον αφορά λοιπόν τα απενεργοποιημένα όπλα. Η πρότασή μου είναι ότι όταν πρόκειται για ένα πυροβολό όπλο το οποίο έχει τροποποιηθεί για να μπορεί να ρίχνει μόνο άσφαιρα, ε, ναι, ε, τότε θα πρέπει να το συνεχίζουμε να το θεωρούμε πυροβόλο όπλο. Να μην περνάει στην κατηγορία ε, Β. Όσον αφορά τα επενεργοποιημένα, θα πρέπει να θεωρούνται πραγματικά επενεργοποιημένα μόνο όταν η διαδικασία δεν μπορεί να αναστραφεί. Μόνο όταν είμαστε σίγουροι ότι το όπλο δεν μπορεί πια να ξαναχρησιμοποιηθεί. Με πραγματικά πειρά. Και η νέα νομοθεσία ευρωπαϊκή για την απενεργοποίηση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, αλλά έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει τεχνικές ελλείψεις, έχει δημιουργήσει ανησυχία σε πολίτες οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν την νομοθεσία, να τηρήσουν την νομοθεσία, αλλά δεν μπορούν ακριβώς εξαιτία αυτών των τεχνικών προβλημάτων της και αυτό έχει και επιπτώσεις στην δημόσια τάξη. Γι' αυτό έχω αποβάλει την πρόταση να, με τεχνική τροπολογία να επανεξετάσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν αποτελούν πυροβολά όπλα. Ε, και είναι τα όπλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να αποστέλουν μηνύματα συναγερμού ε, για φωτοβολίδες κτλ. Ε, αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με τα πυροβολά όπλα. Το ίδιο για τις ρέπλικες. Εάν, εκτός εάν ε, συμπεριλαμβάνουν ένα ουσιώδες εξάρτημα του όπλου. Το κατά πόσον λοιπόν θα συμπεριλαμβάνει ένα ουσιώδε εξάρτημα του όπλου είναι αυτό που θα μα επιτρέπει να αποφασίζουμε ξεκάθαρα εάν πρόκειται για πυροβόλο όπλο ή όχι. Έχω, έχω μάθει ότι ίσως να μην είναι νομικά απαραίτητο να υπάρχει σήμανση σε κάθε ένα από τα ουσιώδη εξαρτήματα. Τώρα θα ζητήσω περισσότερες διευκρινήσεις για να καταλήξουμε στο πιο ακριβό, ποια ακριβώς από τα ουσιώδη εξαρτήματα των όπλων θα πρέπει να φέρουν σήμανση. Όσον αφορά τώρα την ανταλλαγή πληροφοριών, είναι πολύ σημαντικό να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται οι αρχές επιβολές του νόμου και να τις ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ίσως χρειαστεί να υποβάλω νέες ε, τροπολογίες έτσι ώστε να καλυφθούν τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και με βάση την συζήτηση που θα έχω σήμερα με τους εκπροσώπους της ε, Europol. Θα συμπεριλάβω λοιπόν ε, κάποιες προτεραιότητες προτάσεις για το πώς θα πρέπει να γίνεται η κοινοποίηση όταν κάποιος αγοράζει όπλα. Γνωρίζω ότι οι γαλλικές αρχές ε, και άλλες αρχές κρατών μελών ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, όσον αφορά την αποθήκευση, κάποια κρατημέλη ε, ζητούν να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση στις προδιαγραφές για την αποθήκευση όσον αφορά για τις, τις ε, ε ιατρικές ε, εξετάσεις των κατόχων. Ε, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να ε, επαφίεται στα κράτη-μέλη, αλλά κάθε κράτος μέλος οφείλει να έχει μια τέτοια διαδικασία. Όσον αφορά τις πωλήσει μέσω ίντερνετ. Θα επιτρέπονται, αλλά η τελική παράδοση του όπλου θα γίνεται με φυσική παρουσία του αγοραστή έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται ότι εκείνος που τελικά αποκτά το όπλο έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τη δυνατότητα να το αγοράσει. Όσον αφορά τώρα τα πυρομαχικά, σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ε, εξαιρέσεων όταν κάποιο κράτο μέλο θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει στην κατοχή του ένα πυροβολόπλο υπό ε, ξεχωριστέ υποφυσιολογικέ συνθήκε. Δεν θα μπορούσε για λόγου μελέτη, για λόγου ε, δημόσια ασφάλεια στι αρχέ του, για παράδειγμα, και ε, θα προτείνω να υπάρξει μια συγκεκριμένη εξαίρεση στο άρθρο 6, βέβαια με τη ρήτρα ότι αυτή δεν θα πρέπει να δημιουργεί κινδύνου για τη δημόσια ταξική ασφάλεια. και βεβαίως θα δίνεται και η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εξετάζουν και να διασφαλίζουν ότι δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια, ιδίω όταν πρόκειται για την αποθήκευση ενός όπλου σε ένα χώρο όπως ένα μουσείο ή μια προσωπική συλλογή. Τώρα, η χρήση, μάλλον το να τοποθετήσουμε αντικείμενα τα οποία προσυδειάζουν σε όπλα στην κατηγορία Α θα είχε δημιουργήσει πολλά νομικά προβλήματα. Για παράδειγμα γνωρίζω ότι στη Γερμανία αυτό δεν θα ήταν ε, εφικτό και γι' αυτόν τον λόγο θα προτείνω μια τροπολογία για το άρθρο 7 έτσι ώστε να καλέπτονται μόνο τα αυτόματα όπλα τα οποία έχουν μετατραπεί σε αυτόματα. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο αν έχετε προτάσει θα με βοηθούσατε. Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά αυτά τα πυροβόλα όπλα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο ορισμός της κατηγορίας Α θα είναι επαρκώς ευρύς για να επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές να επιτελούν το έργο τους, αλλά ταυτόχρονα να μην δημιουργήσουν και πρόβλημα με την νομική τάξη κάποιων χωρών. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει κάνει μια πρόταση όσον αφορά τις μετατροπές που υπάρχουν κάποιες ανησυχίες εδώ όταν γίνεται μια μετατροπή η οποία δεν είναι ουσιώδης, για παράδειγμα από, ε, στο, στο γεμιστήρα. διευκρίνηση, η νομοθεσία δεν καλύπτει ε, Αντίκε, παλιά όπλα, δηλαδή αν έχετε κάποιο του φέκη του προηγούμενου αιώνα δεν θα χρειάζεται να εφαρμόσετε τη σήμανση. Θα προσπαθήσω επίσης να βρω περισσότερες διευκρινήσεις για αυτές τις μετατροπές. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό με το σύστημα το ηλεκτρονικό για την υποβολή των, τροπολογιών. Γι' αυτό θα προτείνω να παραταθεί μέχρι την επόμενη Πέμπτη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Γι' αυτό σας προτείνω να στείλετε τις τροπολογίες σας μέχρι την επόμενη Πέμπτη 12 το μεσημέρι, εάν δεν έχει πρόβλημα και γραμματεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε σωστές διατυπώσεις, να είναι οι τροπολογίες κατάλληλα διατυπωμένες, μη βιαστούμε χωρίς λόγο. Γνωρίζω ότι αυτά τα θέματα συζητούνται ευ... ευρύτατα στα κράτη-μέλη. Στο Συμβούλιο υπάρχουν και πολλές ομάδες εργασίας και πολλές τεχνικές ομάδες εργασίας που ασχολούνται με αυτά. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τώρα αρχίζουμε τις παρεμβάσεις των σκιωδών. Πρώτη, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Βίκη, πολύ καλή η εκθεσή σου. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους εμπειρογνώμες μας βοήθησαν με τα ε, τεχνικά σημεία για να πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των ε, πολιτών και να μην έχουμε όμως ε, γραφειοκρατία αχρίαστη και περιορισμούς αχρίαστου. Οπότε, για να δούμε τώρα τα μέρος ζητήματα το οποίο μας είπες Βίκη. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα και τη σχετική κατηγορία, εγώ συμφωνώ ότι ε, στην αρχή το σχέδιο του κειμένου ήταν πάρα πολύ ασαφέ αυτό που προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για για τις διάφορες κατηγορίες, για τις ε, τα ημιαυτόματα, το α7 και επομένω νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να μείνει το κείμενο όπως λες εσύ και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις απομιμήσεις γιατί προς το πάνω έχουμε βρει πιστικά επιχειρήματα που να έχουν προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ασφάλεια εάν επαναδιατυπώσουμε τις κατηγορίες. Τώρα όσον αφορά τα ουσιώδη εξαρτήματα και την επισήμανση Επίση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει ε, δυνατότητα ανείχνευση και να υπάρχει κάποιο σύστημα μαρκαρίσματο, α το πούμε, σημαδεύονται. Αλλά δεν μπορούμε να σημαδεύσουμε βέβαια όλα τα ε, κομμάτια του όπλου, όλα τα εξαρτήματα, αλλά να εναρμονίσουμε το σχετικό πρωτόκολλο και επίσης συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά το ότι θα πρέπει τα ουσιώδη εξαρτήματα να σημαδεύονται και όταν αυτό είναι εφικτό να είναι δηλαδή ρεαλιστική η προσέγγιση στην ε, ε η τροπολογία 25 μας λες τι γίνεται με τη θέση που είναι ο γεμιστήρας αλλά είπαμε πριν να δούμε τώρα κατά πόσο θα γίνει κάποια διάκριση πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το ποια κομμάτια του όπλου θα ε, σημαδευτούν. Έχουμε βέβαια και το θέμα των ιατρικών ελέγχων. Θα πρέπει κάποιο να είναι σωματικά ή ψυχικά. Ε, μπορεί να κατέχει ένα όπλο. Και συμφωνώ εκεί που είπε ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα ισχύοντα συστήματα στα κρατημέλη. Σε κάποια κρατημέλη ήδη υπάρχουν κάποιοι δόκιμοι τρόποι εξέταση. Ε, δηλαδή την ευθύνη αναλαμβάνει ένα ιατρός ο οποίος ε, αναφέρει σχετικός εάν ο ε, ασθενής δεν είναι εις θέση να κατέχει όπλο. Και, όπως είπε στην τροπολογία, θα πρέπει να υπάρχει ένα στεγανό σύστημα ελέγχων στα κράτη-μέλη. Το θέμα τώρα ε, των, της διάρκειας, της χρονικής της άδεια οπλοφορίας, τώρα να την κάνουμε πενταετή, για να δούμε στην Σουηδία έχουμε 700.000 ε, άδειε οπλοφορία και καλύπτουν 2 εκατομμύρια όπλα. Αυτό όμως μας δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατία. Ε, μας λένε οι αρχές ότι πρόκειται για πολύ μακρά διαδικασία και σωρεύεται αδικπεραίωτη ότι Οπότε θα πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα υπάρχει καταπολέμηση της παράνομης πώλησης όπλων και διακίνησης και όλα αυτά, αλλά και διασφάλεια. Άρα πώς να δούμε πώς θα εκεί θα κάνουμε και όχι όσον να περικόψουν τη διάρκεια της άδεια. Επίσης λέμε εδώ πέρα για την ασφαλή αποθήκευση ε, γιατί οι πολίτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όπλο για αθλητισμό, για κάποιους ε, τελείως νόμιμους ε, τρόπους θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση στα όπλα ή αυτοί που δεν τα χρησιμοποιήσουν για κακό σκοπό. Άρα ε, σωστά τα λέει το κείμενο. Τώρα όσον αφορά τις πωλήσει εξ θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια αλλά να είναι αναλογική η ρύθμιση γιατί έχουμε και αυτούς που μένουν στην ύπεθρο. Άρα να προβλέπονται οι πωλήσει εξ και να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της άδεια και από την αστυνομία ε, και από τον πολιτή αλλά τώρα στο, στο, στο μέσο του πουθενά στην Λαπωνία πώς να γίνουν όλα αυτά δεν γίνει με την τελευταία φάση της διαδικασίας πώλησης ε, και, και αμφιβάλλω αν προσθέτει και ασφάλεια στο σύστημα Άρα να μην υπάρξει απαγόρευση των πωλήσεων εξ αποστάσεως. Το τελευταίο είναι σημαντικό που μας είπες, δηλαδή όσον αφορά ε, το να ε, κοινοποιούνται οι πληροφορίες, άρα θα πρέπει να εξονίσουμε την οδηγία ανταλλαγή των αριθμών πρακτικών, διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των κρατών μελών, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε το διαχωρισμό μεταξύ ε, νόμιμης κατοχής όπλων που δεν θα πρέπει να καταλήξουν στα λάθος χέρια. Επίσης ε, προσβλέπουμε και εγώ και άλλοι σχεδοσυγητές στο να συνεχίσουμε την συνεργασία μαζί σου. Νομίζω θα πετύχουμε σωστή ισορροπία. Θα δούμε και τις ε, τροπολογίες που θα κατεβάσουμε και θεωρώ ότι εδώ μας ξεκαθάρισες πολλά σημεία του κειμένου της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που κατά του ΕΛΚ δεν ήταν τόσο σαφή. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν. Και τώρα πάμε στους σοσιαλδημοκράτες και το λόγο έχει ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Βίκη για τη δουλειά τη μέχρι εδώ και ακόμα όμως θα πρέπει να κάνει πολλά για αυτό το δύσκολο θέμα γιατί όπως και η ίδια μας ε, τόνισε το εδώ έχουμε μια περίπλοκη πρόταση αλλά και έχουμε και πολυμορφία του τι ισχύει από χώρα σε χώρα όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία που διαφέρει πάρα πολύ και υπάρχει επίσης ολόκληρη κουλτούρα και παράδοση για το θέμα αυτό, πώς δηλαδή χρησιμοποιούν οι πολίτες τα όπλα πρόκειται για αθλητισμό, για άλλες χρήσεις και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να σταθούμε σε κάποια θέματα που μας είπες και να έχουμε και κάποιες τροπολογίες και να δούμε για ποια συγκεκριμένα σημεία αυτό το, το, το των όπλων. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σημαδεύονται τα όπλα ε, όσον αφορά όλα τους τα σημαντικά εξαρτήματα. Και επομένως να μην μπορεί κανεί να τα λύσει τα όπλα και να, αντικαταστήσει ε, κάποια εξαρτήματα και έτσι να αλλοιωθεί η νόμιμη χρήση. Επίσης είναι πάρα πολύ θετικά αυτά που πρότεινε η δίκη όσον αφορά τα ελάχιστα προπετούμενα, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, όλα αυτά θα αυξήσουν την διαφάνεια Και έτσι επίση παρέχονται κάποιες εγγύσει στον ε, κόσμο, στον κόσμο που θέλει να κάνει νόμιμη χρήση των όπλων. Για να τα χρησιμοποιήσει για διασκέδαση, για χόμπι και όχι για άλλους λόγους. Τώρα όσον αφορά την ε, ιατρική εξέταση, μας ε, προτείνεται την συνεχή παρακολούθηση. Εγώ, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την αρχή τη διαδρομή, δηλαδή την πρώτη εξέταση κατόπιν να δούμε τι είναι το πιο σωστό για τη συνέχεια. Να δούμε τι ταιριάζει στην κάθε χώρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η αρχική προσέγγιση. Εκεί να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, να υπάρχει ομοιογένεια και να υπάρχουν εγγυήσει του ότι το κράτος ε, ε, ξέρει ε, ότι είναι κατάλληλη για όπλο η υγεία πνευματική σωματική αυτού που θέλει να κατέχει όπλο. Τώρα για τα μουσεία και για τις συλλογές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει εδώ μια διάκριση. Άλλο τα μουσεία και άλλο οι, εκλογές, οι συλλογές και οι συλλέκτες. Υπάρχει χώρος στο κάθε μουσείο που έρχονται τα όπλα, τα ε, καταγράφουν και εκτίθενται την ιστορία κλπ. Οι συλλέκτες τώρα είναι κάποια πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, τα οποία συλλέγουν και κατέχουν τα όπλα. Γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ε, ορισμός, νομικός ορισμός για το τι εστί συλλέκτης. Ε, αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από το να κάνουμε αυτή τη διάκριση για την ρύθμιση σχετικά με τα μουσεία και του συλλογέ. Ε, ναι, αντικειμενικά δεν μπορεί το ένας να μπει στα χωράφια του άλλου. Είναι, ας το πούμε, αντικειμενική η κατάσταση στα μουσεία, ενώ τη συλλογή ε, η κατάσταση είναι πιο υποκειμενική. Τώρα να αφορά τις ε, πωλήσει με το ίντερνετ. Ενδιαφέρουσα η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα το είναι επεξεργαστούμε για να καταλήξουμε σε συμβαστική διάταξη και σχετικά με τα πυρομαχικά. Αλλά το πιο λεπτό σημείο είναι αυτό που αφορά την επαλήθευση για πωλήσει, αγορές ε, και ποιος δίνει την άδεια. κρατική αρχή, ποιος ελέγχει Είναι νομίζω πολύ σημαντικό να υπάρχει παρέμβαση κάποιας τρίτης κρατικής βέβαια αρχής η οποία να υποχρεούται να προβεί αυτόν τον έλεγχο της ε, ε νομιμότητα και συμμόρφωση προς τον νόμο τέλο πάντων όσον αφορά την πώληση και την αγορά. Τώρα, το δύσκολο θέμα της κατηγορίας υπαριθμών 7 ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ορισμό για το α και να μην έχουμε εδώ ω κριτήριο την ομοιότητα, την απομίμηση, γιατί αυτό δεν μας βοηθάει, δεν μας δίνει κανένα από τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και συζητήσαμε. Θα πρέπει να βρούμε κάποιους κριτήρια αντικειμενικά. Γιατί η ομοιότητα του ενός όπλου προς το ένα είναι κάτι το αόριστο. Άρα, αντικειμενικά κριτηρία τα οποία μπορούν να μας ε, οδηγήσουν σε έναν ε, περιορισμό ε, του πεδίου εφαρμογή της κατηγορίας ε, Α7. Αντίθετα βέβαια το κριτήριο της ομοιότητας διευρύνει πάρα πολύ το πεδίο ισχύω εφαρμογή του Α7. Δεν λέει πολλά ή δεν λέει τίποτα το ότι κάτι προσωμιάζει με ένα άλλο. Άρα θα πρέπει υπομονετικά να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε κάποια αντικειμενική βάση. Και τελευταίο, όσον αφορά την αποθήκευση κάποιων όπλων που πια δεν χρησιμοποιούνται. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ε, ανιχνευσιμότητας. Δεν υπάρχει επιστροφή. Απλώς έχει υπάρξει κάποια δήλωση. Το θέμα κατά πόσο είναι επαλήθευση; Θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε με ένα ε, κριτήριο το οποίο ε, προβλέπει το, τον έλεγχο και την επαλήθευση. Και έτσι εξασφαλίζεται η ανεκνευσιμότητα της ε, πάυσης λειτουργίας του όπλου. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο πρότεινε σχετικό συμβήκη. Οπότε να δούμε και με τους άλλους και τους ηγητές κάποια από αυτά τα σημεία. Νομίζω ότι υπάρχει θετικό κλίμα, θετική υποδοχή αυτής της ε, έκθεσης. Επομένως νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει πολύ θετικά βήματα. Δίτα Χαράντσοβα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βεκίφορτ για το αρχικό σχέδιο της έκθεσης. Αποτελεί μια εξαιρετική βάση πιστεύω για την δουλειά για το σημαντικό αυτό νομοθέτημα. Λαμβάνω θετικά email από τους Τσέχους πολίτες και χαίρονται που υπάρχει πρόοδος από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλωσορίζουν το γεγονός ότι με προσοχή ακούσατε όλους τους εμπλεκομένου φορείς που εξέφρασαν ανησυχίες για την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Υπάρχουν κάμποσα θέματα τα οποία θα ήθελα να δείξω και πιστεύω ότι επ' αυτών θα πρέπει να υπάρξει ένας πιο καλός συντονισμός προκειμένου το κείμενο της έκθεσης να προσεγγίσει ακόμα περισσότερο το ιδανικό. Υποστηρίζω την πρότασή σας σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση των μη αυτόματων όπλων ή κατηγορίας Β και καλώς ορίζουμε τις προτινόμενες 7 κατηγορίες που θα καταργούσε τα αυτόματα που ε, μοιάζουν με μη αυτόματα. Ξέρουμε ότι ήταν προβληματική αυτή η πρόταση εξ αρχής και πιο πολλά ερωτήματα έθετε παρά Έλληνε. Θα προκαλούσε πολλά πρακτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή. Και ωστόσο υπάρχει μια επιπρόσθετη πρόταση σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση, την ταξινόμηση των όπλων στο κείμενο της Επιτροπής, η Α6, τα ημιαυτόματα τα οποία έχουν μετατραπεί από αυτόματα, τα οποία και θα απαγορεύονταν. Ξέρω ότι στην έκθεσή σας περιλαμβάνετε προτάσεις για τα τροποποιημένα όπλα και την διαδικασία τροποποίησης και συμφωνώ απόλυτα και εδώ πέρα πιστεύω ότι χρειάζεται πιο πολύ διευκρίνηση από δική σας πλευράς. Θα προτείνουμε λοιπόν τροπολογία για το τμήμα αυτό της έκθεσης θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω τι σκέφτεστε για την κατηγορία αυτή. Για τις άλλες διατάξεις, καλώς ορίζω τις προτάσεις σας για τον ορισμό των όπλων, τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία των όπλων σε ό,τι αφορά την ε, της εξαποστάσεως του ε, τους ιδρικούς ελέγχους, τα πυρομαχικά, ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα των κρατών μελών να δίνουν εξαιρέσει για ιδιαίτερε περιπτώσει σε ό,τι αφορά την κατοχή κάποιων κατηγοριών όπλων. Αυτό δεν υπήρχε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι λοιπόν που στο σχέδιο έκθεση σα το ξαναβάλλατε. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τις δημόσιες, ε, τα δημόσια ιδρύματα όπως τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, αλλά και για κάποιες ε, επιχειρήσεις ιδιωτικές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Επίσης, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την ε, κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Θα ήθελα να υπάρχουν και περαιτέρω ε, διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για την άρνηση χορήγησης ε, άδεια κατοχής, Πώς θα λειτουργούσε αυτό στην πράξη και ποια πιστεύετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία της διατάξης αυτής. Και υπάρχουν και διατάξεις για την επισήμανση των όπλων και των συστατικών μέρων. Να υπάρχει ένα μητρό λοιπόν που θα έχει πληροφορίες λεπτομερείς για κάθε όπλο το οποίο παράχτηκε και ε, πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε αυτά να ισχύουν μόνο για όπλα τα οποία παράγονται από την εφαρμογή της οδηγίας και μετά. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας, να ευχαριστήσω και τους κοιόδης και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν, κανένα από την ΚΟΕ, επομένως πάμε τώρα και στους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Βίκη για το εξαιρετικό σας έργο γιατί το θέμα είναι προφανώς ευαίσθητο και ιδιαίτερα ευαίσθητο όπως, το ε, όπως είδαμε κινητοποιούνται και οι πολίτες και από τις δύο πλευρές και από εκείνους που πιστεύουν ότι θα μειωθούν οι προσωπικοί τους, ελευθερία, εκείνους που χρησιμοποιούν τα όπλα για αθλητισμό, για συλλογές και επίσης από εκείνη την πλευρά των πολιτών που ανησυχούν για την ασφάλεια, που ανησυχούν για την αύξηση του λαθρεμπορίου όπλων και πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία που γενικά ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο και την ασφάλεια των πολιτών συνολικά που επίσης ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο. Σας συγχαίρω λοιπόν για την επεξεργασία του θέματος και τις διάφορες ακροάσεις που οργανώσατε. Αυτό βοήθησε για να ξεκαθαρίσει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προσπαθεί να εξομοιώσει τους νομοταγείς πολίτες με τους τρομοκράτες ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκείνους που χρησιμοποιούν τα όπλα για σπορ και τους εγκληματίες αλλά ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτρέψουμε στις αστυνομικέ αρχές να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο ε, ε, όπλων και να μην φτάνουν όπλα σε αυτούς τους τρελούς που τα χρησιμοποιούν για μαζικές τρομοκρατικές ενέργειες. Υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση αυτή, ιδιαίτερα στα ζητήματα που αναφέρονται στον αφορά την αποθήκευση, την καταγγελία ε, τυχόν ύποπτων ε, αγοραπολισιών, την ιατρικούς ελέγχους. Κάποιες λεπτομέρειες θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αλλά σε γενικές γραμμές θέσεις είναι σωστές. Τώρα όσον αφορά τις μετατροπές, θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο κ. Κοφεράτη. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο για το ζήτημα με τις τις ρέπλικες. Βεβαίως, ε, κανείς δεν έχει διάθεση να ε, εξομοιώσει ένα παιχνίδι που μοιάζει με όπλο με ένα όπλο. Αυτό δεν θα ήταν σοβαρό, συγγνώμη για την έκφραση, δεν θα ήταν, ε, εν πάση περιπτώσει, νομική απόψεω κάτι που μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Το πρόβλημα όμω είναι με, κάτι με κάποια άλλα αντικείμενα τα οποία μπορούν με μικρέ τεχνικέ τροποποιήσει να χρησιμοποιηθούν ω όπλα, να μετατραπούν σε όπλα. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Έχω επίσης κάποιε απορίε σε σχέση με τα απενεργοποιημένα όπλα, αφού υπάρχει μια νέα νομοθεσία η οποία τα ορίζει. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η νομοθεσία θα έπρεπε να εφαρμόζεται και στα παλαιότερα και στα νεότερα όπλα. Δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Όσον αφορά τώρα ε, τους συλλέκτες, όχι συγγνώμη, τις, τις, τις, ε, ε, τους πολίτες οι οποίοι έχουν όπλα και στους οποίους θα έπρεπε και μπορούμε να ε, επιβάλλουμε τους κανόνες για τον έλεγχο της οπλοκατοχής χωρίς αυτό να δημιουργήσει προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις, στους εθνοφύλακες. Τώρα, να αφορά τους ε, ανήλικους, εδώ βεβαίως και πρέπει να, να, να, να ξεχωριστοί κανόνες, βεβαίως δεν μπορούμε να τους εξοποιώσουμε με τους ενήλικες, βεβαίως ένα όπλο δεν είναι ένα κατάλληλο δώρο για ένα παιδί, Συμφωνώ επίση με τον συνάδελφο Κομφεράτη όσον αφορά τη διάκριση που έκανε ανάμεσα στα μουσεία και τους ε, ε, προσωπικούς συλλέκτες. Εγώ θυμάμαι ότι στην ε, επίθεση στο Μομπελιέ είχαν χρησιμοποιηθεί όπλα από, έναν, από μια προσωπική συλλογή. Γνωρίζουμε ότι τα ε, μουσεία έχουν ε, κανόνες ασφαλείας και επιτήρηση πολύ αυστηρότερη και οργανωμένη από ότι ένας συλλέκτης. Επομένως, πρέπει να είναι διαφορετικοί. Εγώ έχω επίσης ένα πρόβλημα, μια απορία σε σχέση με τα αυτόματα που μπορούν να μετατραπούν σε αυτόματα. Μας λένε ότι είναι δύσκολο να δώσουμε ορισμό. Και οι αστυνομικές αρχές από την άλλη μας λένε ότι είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το πρόβλημά τους με συγκεκριμένα είδη όπλων, καλάσνικοφ και άλλα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε στο ίντερνετ και κυρίως από τις ΗΠΑ προέρχονται και εύκολα να τα μετατρέψουμε σε αυτόματα. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί πολύ. Ξέρω ότι κάποιοι θα προτιμούσα να μην αλλάξει η κατηγοριοποίηση των ημιαυτόματων, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε το θέμα και να μπούμε σε περισσότερο βάθο, αφού μα λένε οι ίδιε αστυνομικέ αρχές ότι έχουν πρόβλημα με αυτά τα όπλα. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για το έργο σας μέχρι τώρα ε, και αναμένω την επόμενη συνάντηση των σκιωδών για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερα στα θέματα που μας απασχολούν και να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Δεν είναι κανείς εδώ από το EFDD. Αλλά όμως από την ENF έχουμε την κυρία Τροσίνσκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Φόρντι για το έργο σας. Καλύπτεται εν μέρη αυτά τα οποία θέλουν οι συμπολίτε μας η πρώτη τροπολογία μας ε, και θέλουμε να περάσει ότι οι περισσότερες τροπολογία σας αφορούν διάφορες επαφές που και εμείς είχαμε με τους πολίτες και κυρίως με κάποιο είδους ε, κυνηγού, συλλέκτες και άλλους φορείς. Αφήνεται τη διακρατική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη για εξετάσεις, για αποθήκευση Αυτά τα πούμε και στην επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά τώρα τους συλλέκτες, συμφωνούμε με την τροπολογία σας παρθμών 14. Οι ισχυρισμοί της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι είναι βάσιμοι και παράλογοι. Και στην περίπτωση της Τούλου, εκεί έχουμε έναν συλλέκτη ιδιώτη, αλλά ήρθαμε σε επαφή μαζί του και μας είπε ότι τον διαρρήξανε. Τώρα, ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το θέμα της ε, απόδοσης ευθύνη. Ε, επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί η έννοια του μεσίτη του ενδιάμεσου. Αυτός δηλαδή που φέρνει σε επαφή τον αγοραστή με τον πολιτή. Θα πρέπει αυτός να φέρει κάποια ευθύνη όπου δεν προβλέπεται. Από μια μεριά, συμφωνώ με το 4β όσον αφορά του ενδιάμεσου και του κατασκευαστέ όπλων. Τώρα, όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα των όπλων, πρώτα-πρώτα και την πρωτοκόλλησή του σε ένα μητρό. Ε, ε, Ευθύ εξ αρχή υπάρχει ένα πρόβλημα, ίσω όχι για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει πρόβλημα στη Γαλλία, διότι είχαμε κάποιε επαφέ και μα είπαν ότι τα σχετικά μητρό αρχεία ε, δύσκολα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί εκεί έχουν ε, γίνει πάρα, πάρα πολλά λάθη. Και δεν τα λέει αυτό το εθνικό μέτωπο, εμείς. Το λένε οι ειδικοί. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστά μήτρα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα πυροβολόπλα. και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Θα πρέπει να εργαστούμε για να το ξεκαθαρίσουμε στην έκθεσή σας. Τώρα όσον αφορά την αγορά από το Ιντερνετ, τροπολογία 21, ρεαλιστικά τα λέτε, αλλά βέβαια υπάρχει το αντίφαση. Γιατί έτσι δεν γίνεται παράδοση στα, χέρια του αγοραστή από του πολίτη. Επιτρέπεται από τι εθνικέ αλλά δεν λέτε ακριβώ δεν δείχνετε τον τόπο πωλήσεω και αγοράς. Εσείς υποθέτετε ότι όλα αυτά γίνονται στην ίδια χώρα. Αλλά τι γίνεται όταν έχουμε διασυνοριακή συναλλαγή ή και με τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης. Τώρα όσον αφορά το μαρκάρισμα των όπλων θα πρέπει όλα, ε, λέμε εδώ πέρα, θα πρέπει με τρόπο να μπορέσουν να σβηστούν να τα σημαντικά εξαρτήματα και ο συριακός αριθμός ε, όμως είπαμε ότι είναι δυνατόν ε, το, το περίβλημα του όπλου να είναι αποπλαστικό όπως σε κάποια περίστοφα, άρα δεν γίνεται. Εκεί πέρα δεν μπορεί να μπει το, το, το, το σημάδι, αλλά επίσης και σε κάποια ιστορικά παλιά όπλα, αρχαία όπλα, αν το κάνουμε αυτό θα τα καταστρέψουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις συλλογές. Συμφωνούμε πάντως με το 77, την τροπολογία, για το α6. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει τα αυτόματα και τα ημιαυτόματα θα ήθελα να το βάλετε στη, αυτή την κατηγορία γι' αυτά είναι πάρα πολύ δημοφιλή τα όπλα για τους σκόπευτες σε πολλά κρατημέλη οπότε θα πρέπει να ποινικοποιείται ο χρήστης ούτε πρέπει να βλέξουμε με θέματα κατάσχεσης από πλευράς του κράτους σας προτείνουμε επομένω κάποιες τροπολογίες για αυτά που σας μίλησα και κάποια άλλα θέματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Απάντως θα πρέπει να καταπονήσουν το λαθρεμπόριο όπλων και θα πρέπει να αποφύγουμε να γίνουν και άλλες τρομοκρατικές ε, επιθέσεις στην ε, Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Οπότε θα ε, πρέπει να ξεχνούμε ότι κάποιος Ισλαμιστής ή κάποιος μαφιόζος μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το πλαίσιο γιατί άλλωστε είναι διάτριτα τα σύνορα στην Ευρώπη. Έχουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων. Το έχουμε πει αυτά με του ειδικού. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για το εμπόριο και πώ θα μπορούμε να περιορίσουμε ε, τι περιπτώσει των επιθέσεων. Τελειώσαμε, λέει ο πρόεδρο, τον γύρο τραπέζης για του σκιώδες ηγητέ και τώρα έχουμε 12 ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει τον λόγο να είμαι θα πειθαρχημένη γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Άρα είμαι υποχρεωμένος να σας περιορίσω στο ένα λεπτό. Γιατί κατόπιν να πάρει το λόγο η Επιτροπή, αλλά και η εισηγήτρια. Έτσι. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να μιλήσω παραπάνω, αλλά υπάρχει και τεχνικά ζητήματα τα οποία ε, θα τα θέσω στα αγγλικά. Χαιρόμαστε που κινείται η διέκθεση, προ τη σωστή κατεύθυνση. Η διαγραφή οποιασδήποτε σύνδεση μεταξύ τη τρομοκρατία και των νόμιμων αποκατόχων και η αφαίρεση στην αναφορά στου συλλέκτε ω πηγή για την εμπορία όπλων είναι σαφές παράδειγμα και θα πρέπει να σχολιάσουμε και να επενέσουμε την ε, τάση προς την επικουρικότητα στο άρθρο 5 σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, παρακολούθηση, σε ό,τι αφορά τα ιατρικά τεστ, τις ιατρικές εξετάσεις. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο. Ευχαριστούμε την κυρία Φόρτ που ήταν ε, πραγματικά άκουσε τους Μαλτέζους εμπλεκομένους φορείς και επίσης σε ό,τι αφορά τα συστατικά μέρη θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τεχνικές προδιαγραφές για να μην υπάρχουν παραμηνίες. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τους, ε, την μετατροπή και θα πρέπει να τα ορίσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος, η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με του προηγούμενου ομιλητέ. Να συγχαρώ τη Βίκη. Πάρα πολύ ισορροπημένη η έκταση και πολλή δουλειά έκανα, αλλά πολλή δουλειά είχαμε, είχαμε να κάνουμε γιατί υπάρχουν και πολλά συμφέροντα. Θα επικεντρωθώ στο θέμα των συλλέκτων. Οι συλλέκτε πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή και για τον απλό λόγο ότι αν το πεδίο εφαρμογή τη έκθεση αυτή, όπω συμφωνούμε όλοι, είναι να εξισορροπήσει την ε, δημόσια ασφάλεια και την διαθεσιμότητα όπλων, το ότι συνδέεται το θέμα των το συνδέονται οι συλλέκτε με τι τρομοκρατικέ επιθέσει δεν είναι ισορροπημένο. Οι συλλέκτε, τα μικρά μουσεία, θεωρώ ότι θα πρέπει να οριστούν καλύτερα ως όρος. Ενδεχομένω να χρειάζονται και αυτή άδεια για να υπάρχει καλύτερο έλεγχο. Είναι σημαντικό όμως να μην μπουν στο ίδιο καλάθι με τους τρομοκράτες σε ό,τι αφορά τις ε, αγορά στο διαδίκτυο να μην κάνουμε διακριτική να μην προβούμε σε διακριτική μεταχείριση των νησιωτικών χωρών γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν να προμηθεύονται τα όπλα τους και αυτό ελέγχεται έχετε όπως και στη Μάλτα από τις αστυνομικές αρχές είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Φόρτ για την καλή δουλειά που έκανε. Υπάρχουν ωστόσο κάποια σημεία όπου θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποιε λεπτομέρειε. Σωστά απορρίψετε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απο... κάποια ενιαυτόματα, τη νέα κατηγορία Α7, βάσει τη εμφάνισή του αλλά και την α6 την κατηγορία θα πρέπει να την απορρίψουμε ή μία αυτόματα όπλα τα οποία έχουν μετατραπεί από αυτόματα έχουν υποστη μετατροπή αυτή η α, απαγόρευση θα έχει σοβαρές συνέπειες για τους ε, κατόχους τέτοιων όπλων και σε ό,τι αφορά την ε, διάκριση των όπλων αυτών. Στην τροπολογία 13, ότι οι συλλέκτες θα μπορούν να, μπορούν να κρατάνε τα όπλα κατηγορίας Α5. Σωστό, αλλά δεν επαρκεί. Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα και αγοραπολασία τέτοιων όπλων. Και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τα υποχρεωτικά χρονικά όρια για την απλοκατοχή, γιατί θεωρώ ότι αυτό αυξάνει μόνο την γραφειοκρατία και την αβεβαιότητα και όχι την ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Κάρας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια αλλά και τους συναδέλφους. για την αντικειμενική συζήτηση που γίνεται. Γιατί ε, κοιτώντας ε, κάποιες... Ε, ανακοινώσει τύπου και κάποια πράγματα που γράφονται στα μέσα ενημέρωση, βλέπω ότι συχνά χρησιμοποιούν αυτή την οδηγία για να ρίξουν λάσπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε πιο αντικειμενική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε πολύ η συγγετρία. Και θα ήθελα να πω με πάσα σαφήνεια ότι αυτή η οδηγία ξεκαθαρίζει ότι οι νόμιμοι κάτοχοι όπλων αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της εγκληματική ε, κατάχρησης και της νόμιμης χρήσης. Και εδώ βάζουμε λοιπόν στο επίκεντρο τα χαρακτηριστικά και όχι την εμφάνιση του όπλου. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Ρούμπιχ γιατί Έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, είναι διαφορετικές οι εμπειρίες μας, οι ομοθεσίες μας και η η συγγήτρια το υπογράμμισε αυτό, ότι αυτές τις διαφορές θα πρέπει να τις εξετάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε συστήματα αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα χρειαζόμαστε και φυσικά θα καταθέσουμε και τροπολογίες και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αλλαγή της προσθεσμίας για την κατάθεση των τροπολογιών. Ο κύριος Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που μόλις είπε ο συναδελφός Κάρας. Κοιτώντα αυτά που μου λένε οι πολίτες από την περιφερειά μου κάθε εβδομάδα. Μου λένε, μα τι σκεφτόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κατέθεσε την πρόταση. Και κοιτώντα αυτά που είπε και η Κουράτσα Μπίλτη, συνάδελφο και η συγγήτρια, ε, θεωρώ ότι όχι μόνο δίνουμε μια αντικειμενική διάσταση, αλλά επικεντρωνόμαστε και επί των ουσιωδών σημείων. Πώς μπορούμε να δώσουμε μια, ένα ενιαίο χαρακτήρα στην οπλοκατοχή στην Ευρώπη, προκειμένου παντού να έχουμε τα ίδια πρότυπα ασφαλείας. Σίγουρα είναι μια επιτακτική ανάγκη, ανεξάρτητα από τις, επιθετικές, από τις τρομακτικές επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, που δίνουν πάντα φυσικά νέα πνοή στο, στις εργασίες αυτές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις άδειε οπλοκατοχής θα πρέπει να μείνουν όπως έχουν στα κατημέλη σήμερα και θα πρέπει να κοιτάξουμε τις προτινόμενες κατηγορίες χωρίς ωστόσο ε, να δώσουμε, να, κάνουμε, να βάλουμε σε μνηκτική θέση όλους όσοι έχουν αποκτήσει όπλα με νόμιμο τρόπο. Ευχαριστώ και για την επικοδομητική συνεργασία. Σας... E το λόγο. Παρακαλώ, έχεις το Α, συγγνώμη, λάβει το ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα με την εισηγήτρια είχε δύσκολο έργο γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ καυτό και βέβαια δεν πρέπει να εξομοιώνουμε τους τρομοκράτες με τους αυτούς αρέσει να κάνουν σκοποβολία αλλά ε, το θέμα είναι ότι ε, υπάρχουν διάβλοι μεταξύ νόμιμης και παράνομης ε, αγοράς όπλων συμφωνούμε σε πολλά σημεία κύριε Συγγήτρια, αλλά τέλος πάντων θέλω να σας πω σε ποια σημεία θέλω κάποιες διευκρινήσεις, κάποια σημεία που μας δυσκολεύουν ο ορισμός του πυροβόλου όπλου θα πρέπει να συζητήσουμε τα βασικά θέματα και τα βασικά στοιχεία και νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση. Επίσης είναι κάπως αόριστο το, το θέμα, η λύση που δίνεται για τις ε, ιατρικές εξετάσεις. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στο πώς θα γίνει. Για α και β κατηγορία ε, συμφωνούμε, η ομοιότητα ε, επίσης συμφωνούμε ότι δεν είναι τόσο σωστό και θα πρέπει επομένως εδώ να υπάρξει διευκρίνηση και έχουμε περισσότερα προβλήματα με τη, κάποιες προτάσεις σας, δηλαδή την απόρριψη του σχεδίου κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί το κείμενο, όχι να απορριφθεί. Τροπολογία 12. Μας λέτε τώρα ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, κατοχής όπλου κατηγορίας Α ή Β αυτό. Αυτό δύσκολο να το δεχτούμε επίσης και η εξομοίωση συλλεκτών με μουσείων. Προβληματικά σημεία. Και συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε για τους ε, ανηλίκους. Εκεί θα πρέπει να πλαισιώσουμε το θέμα και να μην είναι τόσο ευρύτατες οι διατυπώσεις. Κύριε Γκραπίνη, πολύ σημαντική η έκθεση. Λέγουμε ότι όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και η συγγήτρια ασχολήθηκαν εις βάθος με το θέμα και ο κύριος Κάρας ότι τώρα θα πρέπει να τα πούμε στον κόσμο. Είναι κρίμα να παρεξηγούν τις προσπαθίες μας ο κόσμος. Εμείς δεν θέλουμε να περιορίσουμε τους πολίτες. Το αντίθετο θέλουμε να τους ε, προστατεύσουμε. Θέλω να σας πω τα εξής. Στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής δεν λέγεται τίποτα όσον αφορά την σωματική και πνευματική υγεία κάποιου που θέλει να αποκτήσει πυροβόλο όπλων. Να το λέμε ρητός ότι θα πρέπει να γίνεται ιατρική εξέταση. Άλλο που τα ζήτησα και με την Κομισιόν στο Στρασβούργο. Ότι δηλαδή κάτω των 18 ετών δικαιούνται να έχουν κυνηγετικά όπλα. Απίστευτο αυτό. Δεν το δεχόμεθα αυτό και θα καταθέσω τροπολογία ναι, να κάνουν σκοποβολή, αλλά όχι κυνηγετικά. Τώρα, όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, το τι κάνει κάποιος ανά με το όπλο του, ναι, να το χρησιμοποιεί μόνο αν έχει αδειοπλοφορία. αλλά και να έχει και το πιστοποιητικό καλής υγείας. Θα σας διαβάσω έγγραφα τις προτάσεις μου, αλλά νομίζω θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα όσον αφορά τις ε, ιντερνετικές πωλήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τον ρόλο των ενδιαμέσων που δεν μπορούμε να συλλέξουμε. ελέγξουμε. Ο επόμενος. Η κυρία Σαναλοβά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το έργο της. Πήγαινε η έκθεση προς τη σωστή κατεύθυνση, νομίζω. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα. Όχι αντιπαραγωγικά μέτρα. Δεν έχουμε στόχο να αποτρέψουμε την οπλοκατοχή από εκείνους που έχουν τις, ε, τα απαιτούμενα χέγγια, που είναι σε θέση να κατέχουν όπλο. Βέβαια, ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εκατο, ε, χιλιάδες όπλα που ξεκινούν από την νόμιμη αγορά και φτάνουν στη μαύρη αγορά. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο ε, για την κατηγορία 7 είναι σωστή, αλλά πρέπει να τροποποιήσουμε τη διαδικασία για το 6α. Θα στείλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε κυρία Σενάλογα Ευχαριστώ. Πράγματι λοιπόν πιστεύω εγώ ότι η εκθέση τη κυρία Φόρντ είναι προ σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην τσεχική δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ε, με μεγάλη συζήτηση. Πρωτοφανή μάλιστα συζήτηση ε, για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά ακριβώ αυτό το θέμα των όπλων. Η κατηγορία 7α δεν εμπίπτει πλέον στην οδηγία. Όμως μας δημιουργεί πρόβλημα η κατηγορία 6α. Και ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί περισσότερο το ζήτημα αυτό η κυρία Φόρτ. Όταν γίνεται μια μετατροπή ή μια αυτόματο σε αυτόματο και αυτό δηλώνεται στις αρχές και γίνεται από τον έλεγχο των αρχών, τότε και εφόσον παραμείνει η 6α όσο έχει σήμερα, τότε θα βρεθούν με να πρέπει να επανεξετάσουμε τις περιπτώσεις 40.000 όπλων στην Τσεχία. Και αυτό προφανώς μας ανησυχεί. Γι' αυτό θα προτιμούσαμε να διαγραφεί η πρόβλεψη για την κατηγορία 6α. Τώρα, όσον αφορά τη σήμανση, το εάν θα πρέπει να επισημαίνονται όλα τα ε, εξαρτήματα των όπλων, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να έχει αναδρομική αναεφαρμογή. Ο κ. Ντάλτον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία κατάφερε να συνεργαστεί με ενδιαφερόμενους από όλους τους τομείς, από όλες τις ε, απόψεις. Χαίρομαι για τι τροπολογίε 81 και 85 που εξαιρούν ορισμένε κατηγορίε όπλων και ελπίζω αυτέ να γίνουν δεκτέ από την Επιτροπή μα. Στόχο είναι να μην δημιουργήσουμε ε, υπερβολικό άφθος και στο σύστημα της, ε, του ελέγχου τη οπλοκατοχή Σε γενικέ γραμμέ υποστήριζα τι απόψει τη ε, Επιτροπής. Το πρόβλημά μου όμως κυρίως είναι με τους νομοταγείς κατόχους όπλων ενώ εμείς θα έπρεπε περισσότερο να ασχοληθούμε με την, με την, την αναζήτηση των παράνομων όπλων. Και όταν αυτά τα όπλα ε, ανοιχνεύονται, συχνά δεν ε, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Τα όπλα, τα μη ανοιχνεύσιμα, τα οποία έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν χρησιμοποιούνται για σπορ, αλλά για εγκληματικές ενέργειες. Επομένως, το πρόβλημά μας δεν είναι να δημιουργήσουμε περισσότερους κανόνες για τους νόμιμους κατόχους, αλλά να εστιάσουμε περισσότερο στην παράνομη προκοτοχή. Ο πρόεδρος της Ισπανίας. Θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί κυνηγοί είναι οργισμένοι στη χώρα μας με αυτή τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γιατί αυτό γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω για εμείς πολλά χρόνια λέγουμε θα πρέπει να προσέξουμε τα θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας οπότε δεν είναι εδώ κάποιο τώρα να μας ε, κάνει μαθήματα πάνω στην ασφάλεια από την άλλη μεριά θέλουμε να σας ε, δώσουμε αυτή στην την εμπειρία αλλά θα πρέπει να ε, περιοριστούμε στα αναγκαία όσον αφορά το, το κυνήγι άρα θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Φορ γιατί κατέβαλε τρομερή προσπάθεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο ε, να κάνει όσα έκανε. Ε, και τα έκανε με εμπειρογνωμοσύνη και οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει με κάποια θέματα όπω η ανταλλαγή πληροφοριών. Μα λέει η Γαλλία ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στα Μητρώα. Εμεί δεν έχουμε λάθη. Έχουμε ε, πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία και για του κυνηγού η Guardia Civil, η Εθνοφυλακή ε, είναι πανάφτηρη. Και τι γίνεται λοιπόν με τα όπλα που είναι στα ντουλά Δηλαδή αυτά όλα τα κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και σα ε, ευχαριστώ για αυτή την πρόταση Βίκη γιατί έτσι νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και μαζί με τους ανθρώπους από Γερμανία και Αυστρία να είμαστε σοβαροί. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, και πάλι ευχαριστώ. Συγγνώμη αν υπερεύνει το όριο. Κυρία Γιακοντσάρη, ευχαριστώ πολύ. Θα είναι καθοριστικό το σχέδιο αυτό, γιατί το θέμα είναι να μην εξαπλωθούν τα παράνομα όπλα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Αλλά αυτό προκαλεί προβλήματα και σε εθνικό επίπεδο σε πολλές περιπτώσεις Αυτό λαμβάνεται λοιπόν υπόψη. Είναι σημαντικό το ζήτημα του άρθρου 6 και νομίζω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα γιατί μιλάμε για μια απαλλαγή σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε περίεργες ερμηνείες, ξέρετε, και μπορεί ο κόσμος να ε, δράσει με ακατάλληλο τρόπο. Αν ευχαριστήσω πάρα αυτά την εισηγητρία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και να δώσουμε και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στην εισηγητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας απαντήσω σε ένα-δυο λεπτά και να πω καταρχάς ότι θεωρούμε ότι η έκθεση της κυρίας Φόρτ περιλαμβάνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχουμε και δύο σημεία σημαντικά. Καταρχάς, σε πεδίο της εφαρμογής της οδηγίας, όπως ξέρετε, σε ό,τι αφορά τα μουσεία, έχουμε πει ότι μια ευελιξία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, αλλά σε ό,τι αφορά την ευελιξία αυτή δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε και στους συλλέκτες. Θα πρέπει οι συλλέκτες να συνεχίσουν να έχουν όπλα, αλλά με τους όρους ε, που ε, ισχύουν και για τον αθλητικό κλάδο και τομέα. Θεωρούμε ότι λοιπόν θα πρέπει να υποκριθεί στις ίδιες κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία Α τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν κάποιες εξαιρήσει και διατύπωση στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτη και θα μπορούσε να ισχύσει για διάφορους τρόπους. Άρα οι εξαιρεσει θα έπρεπε να περιοριστούν σε θέματα που άπτονται τη ασφάλεια, όπως για παράδειγμα το θέμα της Φιλανδίας για τους εφέδρους. Για την κατηγορία των όπλων τώρα να σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τα μία αυτόματα γιατί μιλάμε για τα μη αυτόματα τα οποία είναι σε θέση να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές που φτάνουν στην Ευρώπη και πολλούνται για παράδειγμα από τον Ισραηλινό στρατό και την χάνουν μετατραπείς και θεωρούμε ότι αυτά τα όπλα θα πρέπει να περιοριστούν για στρατιωτικές χρήσεις και να χρησιμοποιούνται μόνο από το στρατό και τα τεχνικά κριτήρια θα πρέπει επίσης να δεθούν σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και να δώσουμε τώρα το λόγο στη Δίκη Φόρντ για να, να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά θέλω να απαντήσω και σε κάποια από τα σχόλια τα οποία ακούσαμε. Και συγχωρέστε με και με τη σειρά για τη σειρά απαντήσω. Για τις πωλήσει στο διαδικτύο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τελικό σημείο στο οποίο θα ελέγχεται ποιος αγοράζει. Αν θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εξαίρεση για τις υπαίθριες περιοχές, τις περιοχές στην Υπέτρο, να την προτείνετε παρακαλώ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να μην υπάρχει έλεγχος στις πωλήσει online. Και κοιτώντα και το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πάρα πολύ περιοριστικό. Στις πιο πολλές χώρες λοιπόν υπάρχει τελική επαλήθευση, τελικός έλεγχος για να ελέγξουμε ότι όντως πολλούμε στο άτομο το οποίο μπορεί να αγοράσει και θεωρώ ότι χρήσιμο θα ήταν να γίνουν και άλλες ε, προτάσεις για τη διατύπωση για τα απενεργοποιημένα πυροβολά όπλα και για την ε, παρακολούθηση τους ε, σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε ο Σέτζιο. Σέργιο, δεν νομίζω ότι έτσι επιλύεται το θέμα των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων. Το απλά να μπορούμε να τα παρακολουθούμε και να τα επισημαίνουμε. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες απενεργοποιημένα όπλα τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Ε, υπάρχει πραγματικά σύστημα κλειδώματος το οποίο δεν αναστρέφεται. Και θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια βάση δεδομένων. Γι' αυτό μίλησα για πρότυπα για να διασφαλίσουμε ότι τα πενεργοποιημένα πραγματικά δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Για τα ε, ουσιώδη συστατικά μέρη και την σήμανση. Περίπλοκο το ζήτημα, γιατί ακούσαμε του σοσιαλιστές να μας λένε ότι κάθε ουσιώδες ε, συστατικό μέρη θα πρέπει να επισημάνεται, αλλά ένας Ιταλό κατασκευαστή μας είπε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Θέλω λοιπόν να συλλέξω τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη για να καταλάβω ποια συστατικά μέρη πρέπει να επισημένονται και κατά πόσο η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται και για τα ιστορικά αντικείμενα, τα συλλεκτικά αντικείμενα. Σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία, προσπάθησα να πω ότι, κοιτάξτε, αυτό είναι το μουσείο, αυτό είναι ο συλλέκτης. Και προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να ορίσουμε το μουσείο και το συλλέκτη. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να τα διακρίνουμε απόλυτα, γιατί υπάρχουν υπερβολικά πολλές αλληλεπικαλύψεις και σε κάποιε περιπτώσεις ο συλλέκτης μπορεί να είναι ένα τραστ, ένα καταπίστευμα, να έχει κάποια περιθώριο σύγχυση. Και προσπάθησα λοιπόν να αυξήσω έτσι τον πύχη για όλους όσους κατέχουν ιστορικά τέτοια συλλεκτικά όπλα και να δίνονται περιορισμένες ε, άδειε στα άτομα αυτά, στα ιδρύματα αυτά και να μελετήσουμε το τι ακριβώς κάνουν τα άτομα αυτά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εξαίρεση στο άρθρο 6, δεν αποτελεί αυτό πλήρη εξαίρεση. Ξέρω ότι κάποια μουσεία θα θέλουν να εξαίρεται απόλυτα από το πεδίο εφαρμογή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ανταυτού δίνουμε στα κρατημέλη ε, αυστηρούς περιορισμούς για το ε, ε, σε ποιους θα μπορούσαν να δώσουν τις θερμότητες αυτές. Αυτό είναι μία πρόταση, αλλά όπως σας είπα μπορεί να υπάρξουν και άλλες. Για την ερώτηση της ΔΙΤΑ ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών και το πώς ανταλλάσσουν οι κρατικές αρχές αυτές τις πληροφορίες ιδιαίτερα για το ποιος δεν λαμβάνει ε, άδεια. Γι' αυτό θα συναντηθώ και με τη Europol. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν νομίζω ότι είναι εφικτό για κάποιον που βρίσκεται στη Γαλλία να προσπαθήσει να μπει σε ένα σύστημα ε, και να συνδεθεί με την τσεχική βάση δεδομένων. Θα ήταν τέλειο να μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό πραγματικά λειτουργεί και δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει να περνάει αυτό από κάποια κεντρική αρχή σε κρατικό επίπεδο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε σε αυτό να δω. Για το α6, α7. Να δούμε και άλλες προτάσεις. Καταθέστε και άλλες προτάσεις. Ξέρουμε ότι το... η διατύπωση του α7 δεν λειτουργήσε, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν τους αρέσει και το α6, η Ευρωπαϊκή Ευρωπή έθεσε και το θέμα των Ισραηλινών πυροβόλων όπλων. Και αυτό άλλο ζήτημα. Θα ήθελα να δω όλε τι εναλλακτικέ λύσει που έχουμε στο σημείο αυτό για την επισήμανση και κατά πόσον θα ισχύει η επισήμανση για τα νέα προϊόντα και πάλι είναι τεχνικό το ζήτημα και πιστεύω ότι τα πιο πολλά σύγχρονα πυροβολά όπλα θα είχαν ήδη επισήμανση. αλλά θα πρέπει να λειτουργεί, να είναι σωστή και κατάλληλη η επισήμανση. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ισχύει αυτό και για τις αντίκες και για άτομα τα οποία τα αγοράζουν και συμμετέχουν σε ιστορικές έρευνες. Για το θέμα του ίδιου θεωρώ ότι οι συλλέξτες <coughs> θα πρέπει θεωρώ ότι η τροπολογία επιτρέπει στους συλλέκτες και στα μουσεία να κάνουν αυτό που θέλουν αν έχουν άδεια τύπου άρθρου 6. Αν δεν είναι αυτή η διατύπωση, ενδεχομένως να πρέπει να προτείνουμε κάτι διαφορετικό. Για τους ανηλίκους φαίνεται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να το ψηφίσουμε στη τελική ανάλυση. Αλλά και πάλι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε ποιες ήταν οι απόψεις σας για την αυτοάμυνα. και ίσως θα μπορούσα να το συζητήσω αυτό με τους δύο βουλευτέ που το έθεσα. Στον Ηνωμένο Βασίλειο ξέρω ότι στη Βόρεια Ιρλανδία τα άτομα τα οποία ήταν υπό απειλή και είχαν απειληθεί, σε κάποιες περιπτώσεις είχαν άδεια να φέρουν ένα διαφορετικό είδους ε, όπλα. Και αυτό ισχύει ακόμα και για συναδέλφους μας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους ή για οποιονδήποτε διατείνεται ότι έχει δεχτεί απειλή. Όχι, ε, πρόκειται για πολύ αυστηρές ε, περιπτώσεις, μάλλον για περιπτώσεις με, που είχαν ε, πάρει σχετική άδεια υπό πολύ αυστηρούς όρους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό υπάρχει και ως περίπτωση και σε άλλα κράτη-μέλη για τις ρεπλικές, τα απομιμήσεις οτιδήποτε μπορεί να τύχει μετατροπής και να χρησιμοποιηθεί ως πυροβόλο όπλο σύμφωνα με το άρθρο 1.1 ε, ε, θεωρείται πυροβόλο όπλο. Οτιδήποτε θα μπορούσε να τύχει τέτοιες μετατροπής. Ακόμα, αν είναι μάλλον παιχνίδι και δεν έχει ε, οποιαδήποτε τέτοιο θετικό μέρος, εξαιρείται. Αυτό εννοεί η διατύπωση. Ευχαριστώ. Καλώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρο. Στι τρει τελευταίε συνεχίσουμε τη συνεδρία μα και θέλω να σα υπενθυμίσω για να ολοκληρώσουμε την πρωινή συνεδρίαση ότι